Νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Wir sind zwar noch nicht so zahlreich, aber ich hoffe mal, dass der eine oder die andere vielleicht noch. Δεν ξέρω αν θα προσέλθει κάποιος συνάδελφος ή όχι. Ακόμα, γιατί λείπουν κάποιοι. Αλλά επειδή είναι φορτωμένη για μία ακόμα φορά η μερίσια διάταξή μας για σήμερα, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας ε, καλωσορίζω λοιπόν όλους θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, και ξεκινούμε με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, ε, δηλαδή την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ή αιτήματα για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Σας είχα ήδη ενημερώσει ότι αύριο θα αλλάξει η σειρά των ψηφοφοριών, αύριο το πρωί πάντα. Δηλαδή η ε, γνωμοδότηση διακόνου για την ε, πολιτική συνοχή ε, θα είναι πρώτη και στη συνέχεια θα έχουμε την γνωμοδότηση ό,τι αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε περνάμε στο σημείο 2 τη ημερήσια διάταξη, έγκριση δηλαδή των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 22η και 23η Ιανουαρίου του 2018. Έχετε λάβει αυτά τα πρακτικά στα εγγραφά σα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω να ζητάει και πάλι ε, κανείς το λόγο, οπότε θα ήθελα να σας ε, προτείνω να θεωρήσουμε ως εγκεκριμένα αυτά τα πρακτικά εάν μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Περνάμε στο σημείο 3 της σας διάταξης ανακοινώσεις της Προέδρου. Να σας ενημερώσω λοιπόν ως προς τη Γερμηνία ότι σήμερα έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσέχικα, ε, τονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβένικα, βουλγάρικα και ρουμανικά ως γλώσσες διαρμηνίας. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και web streaming στη σημερινή συνεδρίαση και από εκεί και μετά να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν και αποφάσεις των συντονιστών της 22ης Φεβρουαρίου. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι αποφάσεις ε, της 22ης Φεβρουαρίου που αποστάλησαν την επόμενη μέσω email σε όλα τα μέλη της CULT θα πρέπει να θεωρηθούν πλέον ως εγκεκριμένε αφού μέχρι την καταληκτική προθεσμία της 27ης Φεβρουαρίου δεν ε, υποβλήθηκε κανένα είδου αίτημα για τροποποίηση για διόρθωση. Άρα λοιπόν ολοκληρώνω εδώ και τις ανακοινώσεις από την πλευρά της ε, Προέδρου και περνάμε κατευθείαν στο σημείο 4 της ημερήσια ε, διάταξης, δηλαδή την εξέταση μιας πρότασης νομοδότηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία σύμφωνα με προηγούμενο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17 Μαΐου του 2017. Ε, εγώ η ίδια είμαι εισηγήτρια, οπότε επιτρέψτε μου τώρα να συνεχίσω ως εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πω γνωρίζετε όλοι πω αυτό το σημείο τη σας διάταξη είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό και πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και μια εντελώς διαφορετική διαδικασία την οποία ε, χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και η οποία αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ε, αναφέρομαι δηλαδή στην επωνομαζόμενη διαδικασία του άρθρου 7. Ίσως θα θυμόσαστε ότι το Κοινοβούλιο στις 17 Μαΐου του 2017 είχε υιοθετήσει μια πρόταση ψηφίσματος στο οποίο ε, ζητήθηκε από την Επιτροπή για Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις να συντάξει ε, μια ε, ένα ψήφισμα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή του άρθρου 7 παράγραφος 1 και να υπάρξει το σχετικό αίτημα που θα γίνει προς το Συμβούλιο. Η γνωμοδότηση λοιπόν την οποία σας παρουσιάζω σήμερα εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ίσως να θυμόσαστε επίσης ότι σε εκείνο το ψήφισμα ε, ζητήθηκε από την εκλογική κυβέρνηση να άρει ε, το νέο της ε, νόμο σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με την τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Αυτό το είχαμε ήδη συζητήσει εδώ στη δική μας Επιτροπή και στην συνεδρίαση των συντονιστών είχαμε προσκαλέσει εδώ τον ε, πρίτανη της Central European University, τον κύριο Ιγνάτσιεφ, ο οποίος ε, μας είχε ενημερώσει ε, σε σχέση με την κατάσταση. Και έκτοτε εγώ βρίσκομαι σε επαφή με τον κύριο Ιγνάτσιεφ, έτσι ώστε να ενημερώνομαι ως προς το πού βρίσκονται τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση. Και θα γνωρίζετε βέβαια ότι στο διάμεσο διάστημα και η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά αυτού του νόμου για την τροποποίηση της νομοθεσίας ε, για την τριτοβάθμια, ε, ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αντίκειται στις βασικές ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, εγώ τι τελευταίε εβδομάδε ήρθα και πάλι σε επαφή με τον κύριο Γνάτσεφ, ώστε ακριβώ να ενημερωθώ προς το πού βρίσκονται τα πράγματα, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και μετά από τα όσα μου είπε θα υποβάλω και δύο ακόμα τροπολογίε σε σχέση με αυτή την νομοδοτηση. Και αυτό γιατί μου είχε πει ότι αρχικά είχε προβλεφθεί πω ε, μια ουγγρική αντιπροσωπεία θα μετέβαινε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ προκειμένου να ε, διευκρινιστούν οι σχετικέ ε, διαδικασίε, αλλά η εν λόγω επίσκεψη τελικά ακυρώθηκε από την ουγγρική πλευρά για μετά από τις εκλογές και συγκεκριμένα μία μέρα μετά από τις εκλογές που θα λάβουν χώρα εκεί. Δεν γνωρίζω κατά πόσο πράγματι θα λάβει χώρα μία ημέρα μετά τις εκλογές μια τέτοια επίσκεψη, αν θα παραταθεί περαιτέρω. Πάντως ε, με μια τροπολογία που θα υποβάλω προτείνω να πούμε ακριβώς αυτό το γεγονός ότι δηλαδή ότι λυπούμεθα που η σχετική διαδικασία, η σχετική επίσκεψη ε, αναστέλλεται ξανά και ξανά και δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Έχουμε ήδη στραφεί προς την Ουγγλική κυβέρνηση με την παράκληση να ε, αναζητήσει το ταχύτερο δυνατό μία λύση προκειμένου να διασφαλιστούν και στο μέλλον ή να διασφαλιστεί η συνέχιση της ε, λειτουργίας του Central European University. Αναφέρθηκε από την Ουγγρική πλευρά ότι θα συνεχιστούν οι σχετικέ ε, προσπάθειες προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδο από την Ουγγρική πλευρά και γι' αυτό θεωρώ πω θα πρέπει να το αναφέρουμε μέσα σε αυτήν εδώ τη γνωμοδότηση. Πέραν αυτού, ε, στην γνωμοδότησή μου ε, αναφέρομαι ε, και στο ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης των παιδιών Ρωμά, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα, όχι βέβαια αποκλειστικά μόνο της Ουγγαρίας, αποτελεί ένα πρόβλημα που και άλλες χώρες της ίδιας περιοχής αντιμετωπίζουν, αλλά καθώς αυτό ο κοινωνικό αποκλεισμός στον των περιορίζει ε, την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας και τις σχετικές ευκαιρίες τους, θεωρούμε πως ή θεωρώ μάλλον πω ακόμα και αν δεν αποτελεί αμυγό ουγγρικό φαινόμενο αυτή η διακριτική μεταχείριση του Ρωμά ε, πως καλό θα ήταν να αναφέρεται αυτό το ζήτημα μέσα στην ε, δική μα ομοδότηση. Κάτι ακόμα το οποίο εμπίπτει στο δικό μα τομέα αρμοδιότητα και το, και το οποίο θεωρώ εξίσου ανησυχητικό είναι η ο περιορισμός ε, της ελευθεροτυπίας ε, με βάση εκτεταμένες ε, κρατικές παρεμβάσεις και του αυξημένου κρατικού ελέγχου και νομίζω πως θα θυμόσαστε όλες τις συζητήσεις που είχαμε κάνει σε ό,τι αφορά την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία είχαμε προσπαθήσει να ζητήσουμε από την Ουγγρική πλευρά να αναστείλει κάποιες προτάσεις ε, που είχε κάνει, κάποιε τροποποιήσει ε, προκειμένου ε, μέσω φορολογικών μέτρων να περιορίσει την ανάληψη λειτουργίας αλλοδαπών μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα όπως το Και νομίζω πως αυτό το ζήτημα θα αναφερθεί ιδιαίτερα η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά καθώς αυτό το θέμα αποτελεί και δική μας αρμοδιότητα, θεώρησα σκόπιμο να αναφέρεται στη δική μας γνωμοδότηση, ότι δηλαδή η ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ύψιστο δημοκρατικό αγαθό το οποίο θα πρέπει να τη και τις ανάλογες προστασίας ε, και πρόθεση στην Ουγγαρία. Ε, νομίζω πως ε, στη γνωμοδότησή μας θα πρέπει επίσης να περιοριστούμε μόνο στα ζητήματα εκείνα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας, δηλαδή παιδεία, πολιτισμός, μέσα ενημέρωσης. Ας περιοριστούμε σε αυτά μόνο. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ε, αφήσουμε στη ΛΥΜΠΕ, αλλά και στις υπόλοιπες ε, επιτροπές, ε, καθώς και μια σειρά από περαιτέρω επιτροπές θα τοποθετηθούν σχετικά. Οπότε σας παρακαλώ στις τροπολογίες που θα υποβάλλετε, περιοριστείτε ακριβώς αυτούς τους τομείς αρμοδιότητάς μας. Δεν θα ήταν θετικό, δεν θα δίναμε μια καλή εντύπωση εάν αναφερόμασταν και σε περαιτέρω ζητήματα που δεν αφορούν τη δική μας αρμοδιότητα. Ε, και από εκεί και μετά, βέβαια, επειδή υπάρχουν και σημαντικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις γνωμοδοτήσεις, δηλαδή τον αριθμό των χαρακτήρων, ε, καλό θα ήταν να αναφερθούμε σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τις δικές σα τροπολογίε, τι προτάσει σα, αλλά και τα σχόλια που θα κάνετε τώρα προφορικά στη συζήτησή μας. Να περάσουμε λοιπόν στους ε, σκιώδους ε, εισηγητές. Η κυρία Σόντροβα για το ΕΛΚ κανονικά θα είχε το λόγο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να παρευρεθεί, οπότε δεν ξέρω. Η Σαμπίνα νομίζω θα πάρει το λόγο εκ μέρους της. Ναι, θα διαβάσω εδώ την γραπτή τοποθέτηση της κυρίας Σόντροβα. Αν μου απομείνει χρόνος θα τοποθετηθώ και εγώ μετά, με βάση τη δική μου προσωπική άποψη στη συνέχεια αυτής της παρέμβασης. Η κατάσταση στην Ουγγαρία μας ανησυχεί. Είναι θεμητό να θέτουμε ερωτήσεις και να διαφερόμεθα για την κατάσταση των πανεπιστημίων και των μέσων ημέρας στην Ουγγαρία. Θα πρέπει επίσης να σεβαστούμε και το δικαίωμα της Ουγγαρίας να επιλύει αυτά τα θέματα από μόνη της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προέδρο για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που αντικατοπτρίζει το πόσο σοβαρή εμφανίζεται η κατάσταση στην Ουγγαρία. Σαν ομάδα του ΕΛΚ είμαστε οι πρώτοι που καλούμε περί διαλόγου για, με την Ουγγρική κυβέρνηση για να συζητήσουμε προβληματικά θέματα. Πολλά από αυτά βρίσκονται να εξελίξει και πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρόνο και να δούμε τελικά αποτελέσματα. Το βασικό θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Υπήρξαν πολλές επικρίσεις όσον αφορά την νέα νομοθεσία και αντέδρασε μέσω τροποποίησης του νόμου η κυβέρνηση. αξιολογεί την νομοθεσία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πρέπει να περιμένουμε για την απόφασή του πριν τοποθετηθούμε. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ουγγρική κυβέρνηση να συνεχίσει το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ενδιαφερομένους φορείς και πάντα θα είμαστε προσπιστές της ανεξαρτησίας των πανεπιστημίων και θα τη φωνή μας εναντίον ιαδεσδήποτε απόπειρα που θα ε, καταπιέζει τα πανεπιστήμια για πολιτικούς λόγους. Έχουμε φυλάξει να αφορά τη διατύπωση για την απομόνωση των Ρωμά στα σχολεία, το ΕΛ και είναι υπέρ ίσων ευκαιριών στα σχολεία για όλα τα παιδιά. Η απομόνωση των παιδιών Ρωμά είναι μακροπρόθεσμο δομικό πρόβλημα το οποίο αφορά όχι μόνο την Ουγγαρία αλλά και άλλες χώρες. Οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν λάβει διάφορες συστάσεις επ' αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν βλέπουμε τον επίγοντα χαρακτήρα να αναφέρεται αυτό στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΚΟΛΤ όσον αφορά την ευθερία των μέσων ενημέρωση και την περίπτωση της εφημερίδας Νετσάμτσακ, δεν ξέρω αν την προφέρω σωστά, η κυρία Μπότσκο μπορεί να καλύτερα από μένα, ε, η κατάσταση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Το κλείσιμο της εφημερίδας έγινε από τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, δεν είναι μέσω κυβερνητικής αποφάση. υπάρχουν όμως καταγγελίες που σχετίζεται με το κυβερνητικό κόμμα ιδιοκτήτης. Η κατάσταση δεν απέχει από αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες στην περιοχή, όπως στη Τσεχική Δημοκρατία και στη Σλοβακία. Εν αυτή τη ενία θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μου και προσβλέπω σε καρποφόρες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν η τοποθέτηση κυρία Σόντρουβα. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διακόνου έχει το λόγο. Ε, εν λίνη μάρη, absolut de acord cu propunerea de aviz făcută de... Ε, γενικά ευπρόσδεκτη η άποψη της εισηγήτριας, αλλά έχω ένα σχόλιο σχετικά με όλα αυτά και αφορά το διαδικαστικό. Η διαφορά μεταξύ εκθέσεως και γνωμοδοτήσεως είναι κάτι που αναφέρθηκε από την ε, Πρόεδρο και την εισηγήτρια. Στο κάτω-κάτω μία έκθεση είναι ένας φορέας προς επίτευξη σκοπού. Το ίδιο ισχύει και με γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας. Το πρώτο όμως όχημα είναι με μακροσκελές. Το δεύτερο δεν είναι το μακροσκελέ. Ε, είναι σαν ένα τραμπ. δεν πα και τι βαλίτσε σου μαζί. Ενώ το άλλο είναι τρένο, Φερρυπίν. Ήθελα λοιπόν να συμβάλλω με την άποψή μου και ήθελα να πείσω τους συναδέλφους να μην προσθέσουν πολλά στοιχεία. Ό,τι είναι ασήμαντο να μείνει εκτός να τονίσουμε τα βασικά θέματα, την κεντρική ιδέα. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέλγα Τρούπεν. Σας ευχαριστώ Πέτρα. Ε, ευτυχώς μπορώ να τοποθετηθώ εδώ εκφράζοντας τη δική μου προσωπική άποψη, οπότε να το κάνω. Τώρα, αυτή η περιγραφή μας έκανε στις κατάστασεις στην Ουγγαρία εντάσσεται σε, μια, ε, σε ένα γενικότερο θέμα σε ό,τι αφορά τις διαφορές ανάμεσα στη Δυτική ε, και την Ανατολική, για παράδειγμα Γερμανία, αλλά και άλλες ε, διαφορές. Ένας γνωστός συγγραφέας έγραψε ένα, σύντομο, ε, ε, ένα πρόσφατο βιβλίο ε, ως προς το εδώ στην Ευρώπη και στο ότι δεν έχουμε να κάνουμε με δυτικούς και ανατολικούς και με το γεγονός ότι η πτώση του τείχους και οι πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά την εθνική συνείδηση και τον τονισμό αυτής της εθνικής υπερηφάνειας σε αντίθεση ακριβώς μετά, ε, με την κατάσταση στη Δυτική Γερμανία και την ε, ήττα της ε, από τις συμμαχικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή η εθνική υπερηφάνεια την οποία καταδεικνύουν διάφοροι δεν είναι αυτή την οποία εκφράζουν διάφοροι πρωθυπουργοί και πρόεδροι αυτών των χωρών. Δηλαδή, εάν όλοι δίνουμε έμφαση στην, ε, στη δική μας ε, χώρα, τότε τίποτα δεν θα λειτουργήσει σε επίπεδο ενίσχυσης και εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτά τα λέω εισαγωγικά. Από εκεί και μετά, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπερασπιστούμε με μεγάλη σαφήνεια το κράτος δικαίου και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες. Νομίζω πως η διαδικασία του άρθρου 7 αναφέρεται και σε σχέση με την Πολωνία και είναι σημαντικό πως έγινε αυτό. Γιατί ε, υπόθηκε βέβαια ότι ο Κασίνσκι ή Κασίνσκι για παράδειγμα και ο Ούρμπαν θα εκμεταλλευτούν αυτέ τι διαδικασίε εναντίον του προ όφελό του. Αλλά δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να μην κάνουμε τίποτα. Έχω μία σειρά εγώ για παράδειγμα από φίλου ε, προσωπικού ε, ελεύθερου ε, δημοκράτε οι οποίοι υπερασπίζονται τη δημοκρατία και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των εθνικιστικών κυβερνήσεων και τέτοιων ρευμάτων σκέψη. Άρα λοιπόν όσοι είναι φιλοευρωπαίοι, όσοι επιθυμούν την υπεράσπιση του κράτου δικαίου, όσοι δεν είναι υπέρ του εθνικισμού, όσοι τάσσονται υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, υπέρ του δικαιώματο άμβλωση και ούτω καθεξή, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικά υπερασπίζονται όλοι αυτοί αυτό που βρίσκεται στις, στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις θεμελιώδες μας αξίες. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δασομαστε εμφατικά ε, εδώ να παίρνουμε θέση όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, για ε, ζήτημα θεμελιωδών αξιών, ειδικότερα ως ευρωβουλευτές. Ε, τώρα, αναφέρθηκε ε, σε ό,τι αφορά τους ε, ότι η Επιτροπή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή όχι. Όχι, δεν ισχύει αυτό και θα καταψηφίσω κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεται και ομοφωνία. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, αντιδράσουν, να τοποθετηθούν επί αυτών των γνωμοδοτήσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετικό. Και αυτό που λένε δηλαδή αυτοί οι, ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ε, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ε, διατάζει και επιτάσσει ε, τα όσα εκείνη επιθυμεί με μια προσέγγιση top-down, είναι εσφαλμένα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και ούτε θα ήθελα να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, σε μια χώρα που η Τελωνία, ότι τι θα πρέπει να κάνει σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του κράτου δικαίου, αλλά δεν υπάρχει καμία διαδικασία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εκτελεστικού χαρακτήρα εντολέ στι εθνικέ κυβερνήσει. Δεν είναι τέτοια φύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι λένε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώ δεν, μάλλον ευτυχώ δεν ισχύει. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι απλώ να υπερασπιστούμε εδώ το ευρωπαϊκό ε, πνεύμα. Αυτή λοιπόν είναι βασική μου τοποθέτηση σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα και με αυτό το σκεπτικό θα υποβάλω τι δικέ μου τροπολογίε. Πάντω είμαι βέβαια ότι η δική μα υποχρέωση είναι να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κράτο δικαίου και κατά συνέπεια το κράτο δικαίου σε αυτά τα κράτη-μέλη χωρί καμία διαφοροποίηση των απόψεών μας. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι δεν είναι κάτι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αυτοί υπερψήφισαν τον Brexit ή οτιδήποτε άλλο, θα ήταν εντελώς εσφαλμένο. Ε, δηλαδή, ε, και για την περίπτωση του Brexit, γνωρίζαμε ποιοι είναι εκείνοι που υπερψήφισαν ε, τον Brexit ε, και παρότι σεβόμαστε αυτή την απόφαση, δεν σημαίνει ότι μας βρίσκει σύμφωνος. Σας ευχαριστώ. Έχουν δύο ζητήσει το λόγο, Σβέρ και Μπόσκορ. Και η Σαμπίνε θα πρέπει να φύγει από ό,τι κατάλαβα σύντομα. Οπότε, αν συμφωνείτε να πάρει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να λάβουμε σοβαρές αρμοδιότητες μας στο πλαίσιο της γνωμοδότησης, ε, της έκθεσης ε, της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Και Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ πρόκειται για μια διαδικασία. Όχι για ένα ψήφισμα που μπορεί κανείς να αναφέρει απλά τις απόψεις τους. Θα πρέπει επιμελώς να ελέγξουμε τα πράγματα ε, που είναι κάτι που αντεποκρίνεται στην πραγματικότητα, ε, που υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες κτλ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε πραγματικά στα γεγονότα, στα πραγματικά στοιχεία για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συμφωνήσει βασικές αρχές με την Ουγγαρία και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πολλές φορές ε, έχουμε προβλήματα περισσότερα από ό,τι με άλλες χώρες που έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα, αλλά με το διάλογο και με την επίρρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολλές φορές εκεί που είχαμε ε, να πηγαίνουν τα πράγματα στη λάθος κατεύθυνση διορθώθηκε η πορεία, όπως η ελευθερωτική είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε και έχει φτάσει νομίζω κάπως στα όρια, μέχρι δηλαδή εκεί που μπορούμε να δεχθούμε εμείς από ευρωπαϊκής πλευράς. Δηλαδή η παναχώρηση. Σίγουρα η ελευθεροτυπία πρέπει να δούμε. Ε, υπάρχει πρόβλημα, ε, υπάρχει, υπάρχουν εμπόδια στην ελευθερία του τύπου και θα πρέπει να δούμε και τι επιρροές υπάρχουν από την κυβέρνηση, αν υπάρχουν στοχευμένες στρατηγικές. Θα πρέπει να τα ερευνήσουμε όλα επιμελώς ε, όσα συζητούνται στην έκθεση αυτή και τα σημεία τα οποία άπτονται του άρθρου 7 θα πρέπει να τα δούμε γενικώ κάποιες ε, ανεπάρκειες ή κάποια προβλήματα. Υπάρχουν ε, πράγματα που δεν λειτουργούν καλά στην Ουγγαρία και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα βασικά σημεία, σε συγκεκριμένα σημεία όμως τα οποία άπτονται του άρθρου 7, που είναι οι βασικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Μπόσκορ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν συμφωνώ με διάφορα σημεία και υπάρχουν και κάποια σφάλματα και παρερμηνίες ως την γνωμοδότηση όσον αφορά την παιδεία για τους Ρωμά και τη σχετική νομοθεσία. Ζητώ λοιπόν, συνάδελφοι, να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να στιγματίζετε στην, την Ουγγαρία στην γνωμοδότηση. Ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια κρατών η Ουγγαρία, αντιπροσωπεύει και προστατεύει τις ευρωπαϊκές αξίες και η εθνική κυβέρνηση της Ουγγαρίας ακολουθεί συντηρητικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι η προστασία των γυναικών Απορρίπτων λοιπόν τις κατηγορίες σας που λέτε ότι είναι εθνικιστική η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται αρνητικά το εθνικιστική. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε συντηρητικοί και για μας είναι σημαντικές οι ευρωπαϊκές αξίες. Κάποια στοιχεία της εκθέσεως είναι ασαφή. Φερρυπίν. Δεν αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το ότι οι εθνικές νομοθεσίες στην νότατη εκπαίδευση σε άλλες χώρες μπορεί να είναι πιο περιοριστικές από την αντίστοιχη νομοθεσία της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία έχει κάνει βήματα προς συμβιβαστικές θέσεις. Διαπραγματεύεται. Είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί. Και νομίζω ότι αποδεικνύουμε την προθυμία μας και την καλή μας πίστη και συζητούμε με τους θεσμούς διάφορους φορείς, όπως είναι και πανεπιστήμια στην Κίνα, Φερρυπίν, και το ίδιο μπορεί να γίνει και με το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους εκείνους που είπαν ότι ανάκληση του νόμου δεν είναι κάτι επί καιρό, διότι δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο από το 10 ακόμα. Όσον αφορά την απομόνωση των παιδιών των Ρωμά, είπατε κι εσείς, Πρόεδρε, ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία. Η Ουγγρική κυβέρνηση έκανε πολλά για να αλλάξει την κατάσταση. Τα παιδιά των Ρωμά, Φερρυπίν, από την ηλικία των τριών ετών και πάνω, μπορούν να πάνε σε νηπιαγωγείο και η παρουσία τους στα νηπιαγωγεία έχει αυξηθεί. Οπότε είχαμε θετικά βήματα που έγιναν. Το αναγνωρίζει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ίδια η Επίτροπος, η κυρία Γιουρόβα, είπε ότι έχουν αλλάξει κάποιοι νόμοι σχετικά με αυτό και υπό το φως όλων αυτών των επικρίσεων πρέπει να προβάλλουμε και τα θετικά βήματα πρόοδου και την ανοιχτή στάση της κυβέρνησης για περαιτέρω συνεργασία. Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί τελικά, μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά σημεία αφορούσαν την πολιτική των, για τα μέσα ενημέρωσης της κυβερνήσεως. Να πω ότι το άρθρο 9 του συντάγματός μας λέει ότι προστατεύεται η ελευθεροτυπία και η ποικιλομορφία των απόψεων ε, που εκφράζεται στον τύπο. Και έχουμε νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και ο νόμος λέει ότι οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι έχουν ελευθερία και ό,τι τυπώνεται στα έντυπα μέσα είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους εκδότες και τους ιδιοκτήτες των εφημερίδων. Όσον αφορά την Εύτσα Μουτσακά, αυτή την εφημερίδα και το ότι έκλεισε αυτή η εφημερίδα, αυτό το κλείσιμο δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Η εφημερίδα από το 2007 ήταν ζημιογόνος και ο αυστριακός ιδιοκτήτης το αποφάσισε αυτό. Όσον αφορά την ιστοσελίδα 888.hu, το κλείσιμο αυτό δεν έχει καμία ε, σχέση με την κυβέρνηση. Δεν φέρει ευθύνη η κυβέρνηση. Για το μαύρο κατάλογο των δημοσιογράφων, τη μαύρη λίστα των δημοσιογράφων που δημοσιεύεται εκεί, σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν έχετε πρόβλημα με αυτό, να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο των Μέσων Ενημέρωσης, που είναι ανεξάρτητο συμβούλιο, είναι 9 μελές. Αν διαπιστώσετε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει, μπορείτε να υποβάλλετε σχετική καταγγελία σε αυτό το Συμβούλιο. Δεν σχετίζεται με την κυβέρνηση αυτή στο σελίδα. Δεν έχει καμία ευθύνη η κυβέρνηση. Ε, ελπίζω ότι θα βρούμε συμβιβαστικέ ε, λύσει για να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που είναι δίκαια και αξιόπιστη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Μπόσκορ. Θεωρώ ότι έχει πάρει πολιτική διάσταση ε, το θέμα. Πολλές φορές όμως έχει ε, ξεκαθαριστεί το ζήτημα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν αναφερθεί και οι συμφωνίες με, τις, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία ε, κυρίω ότι τηρεί ε, τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες. Δεν λέει άλλα στη χώρα του και άλλα κάνει. Επίσης ό,τι αφορά αυτό το νόμο περί ανωτά των σχολών. Υπάρχει ένα πρόβλημα ε, για τη μην κατάργηση ακόμη αυτού του νόμου αλλά υπάρχουν και κάποιοι υπενιγμοί και ισχυρισμοί που δεν στέκουν. Εγώ ξέρω την κατάσταση στην Ουγγαρία και δεν είναι τόσο αρνητική όσο ίσως σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο χάρη, άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ε, ε, έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στο θέμα του διαχωρισμού των Ρωμά, το απομόνωση των Ρωμά, των παιδιών από την εκπαίδευση. Μην υπερβάλλουμε λοιπόν. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει εκλεγεί με την πλειοψηφία των Ουγγρών ψηφοφόρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύουν παντού τα ίδια μέτρα και σταθμά και να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάλογα με την περίπτωση. Και άλλου υπάρχουν προβλήματα. Και δεν τα κάναμε τόσο μεγάλο θέμα. αν ε, κλείσει κάποιο σταθμό, κάποια εφημερίδα, κάποιο μέσο τέλο πάντων μαζική ενημέρωση. Ε, Αμέσω ε, ε, οξύνονται τα πράγματα, ενώ μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Αν πρόκειται για την Ουγγαρία για κάποια άλλη χώρα. Πολλές φορές όμως ε, και οι εκλογέ που γίνονται σε άλλες χώρε μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση. Ε, καταλαβαίνω ότι είμαι στη μειοψηφία σε ό,τι αφορά τι απόψει μου πρόεδρο. Από ό,τι ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να τοποθετηθεί. Α, ο κ. Διακόνου θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα θεωρώ ότι είναι σημαντικότατο ακόμα και αναφορά μια γνωμοδότηση. Διότι ίσω δημιουργηθεί προηγούμενο. αυτό είναι ο κίνδυνος. Ακούγοντας τους προλαλήσαντε, σκέφτηκα αυτό που συμβαίνει στη Ρουμανία. Δηλαδή, τηλεοπτικό σταθμός, ένα κανάλι χρεοκόπηση, ήταν χρεοκοπημένο επί πολλά χρόνια. Και κανείς δεν το κλείνει το σταθμό αυτό διότι θα θεωρείται ότι η Ρουμανία περιορίζει την ελευθερία των μέσων. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Πρέπει να το εξετάσουμε από κάθε οπτική γωνία, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ja, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für Ihre... Äh, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις σας. Ανταλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ε, χωρίς αμφιβολία δηλαδή Ένα αμφιλεγόμενο και διαφιλονικούμενο όχι μόνο εδώ στη δική μας Επιτροπή, αλλά στο σύνολο του Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε επίσης πως είναι διαφορετικό το τι αναφέρει ένα σύνταγμα και το τι αναφέρει μια νομοθεσία και διαφορετικό το τι συμβαίνει στην πράξη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, μιας νομοθεσίας. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να υπάρξει ένας νόμος για να περιορίσει για παράδειγμα την ελευθεροτυπία. Υπάρχουν άλλοι μοχλοί άσκησης πίεσης, άλλα μέσα μέσω των οποίων μπορεί κανείς να επιβάλλει περιορισμούς ε, στα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να τους περιορίσει σε τέτοιο βαθμό ε, της, ε, την οικονομική δραστηριότητα που να μην μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να στρέψουμε ε, την ε, προσοχή μας και σε τέτοιου είδους ε, μέτρα, γιατί ο πλουραλισμός, η ελευθεροτυπία, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο ανήκει όχι μόνο στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελεί και κάτι το αμυγός απαραίτητο εγγενώ απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το με ποιον τρόπο περιορίζονται τα δικαιώματα και οι δυνατότητες ε, άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος μέσω διαφορετικών έμεσων δηλαδή τρόπων, όπως ε, για παράδειγμα μέσω φορολογικών νόμων. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η Χέλγα Τρούπελ, ότι δηλαδή πέρα από πατερναλιστικού ε, τύπου ε, συμπεριφορές για τις οποίες κατηγορείται ενίοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αξίες τις οποίες προσυπογράψαμε όλοι και όλα τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της υπογραφής των συνδικών της Ένωσης. Αυτές οι αξίες θα πρέπει να διρούνται όχι μόνο κατά τη χρονική στιγμή ή πριν από την προσχώρηση, για παράδειγμα, της υπογραφής Γιατί θυμάμαι για παράδειγμα το τι είχε συμβεί στην περίπτωση της ε, Κροατίας, πόσο είχαμε πει μην στο γεγονό ότι θα πρέπει να ε, πληρεί όλες αυτές τις θεμελιώδεις αξίες, ότι θα πρέπει να τις στηρεί. Ε, όταν πρόκειται δηλαδή και, μια, για μια χώρα η οποία πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτά θα πληρούνται μέχρι να καταστεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μια χώρα και ακόμα και μετά από την προσχώρηση προφανώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η περαιτέρω τήρηση των λόγω αξιών. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε και σε σχέση με αυτό υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν τηρούνται εν λόγω αξίες ε, όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά μεταξύ διαφόρων χωρών και στην Ουγγαρία στο ένα ή στο άλλο τομέα. Και από εκεί και μετά ναι να πούμε ότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει επιδείξει την πρόθεση να προβεί σε διάλογο. Απλώ αυτό που αναφέρω εγώ στην γνωμοδότησή μου είναι ότι η εν λόγω συζήτηση, ο λόγο διάλογο θα πρέπει να λάβει χώρα με ταχύτητα προκειμένου να διευκρινιστούν το ταχύτερο δυνατό τα πράγματα τόσο για την ε, Central European University όσο και για άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία της στον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια. Ε, αυτή δηλαδή η παρελκυστική τακτική την οποία εφαρμόζει αυτή την περίοδο η κριτική κυβέρνηση δεν είναι αποδεκτικά τη δική μου άποψη εδώ και ένα χρόνο. Και κάτι τέτοιο βέβαια αποβαίνει και εις βάρος της λειτουργίας ε, του ελόγου ε, Πανεπιστημίου της Ουγγαρίας. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να αξιώσουμε από την Ουγγρική κυβέρνηση να ακολουθήσουν μετά από τα όσα μας αναφέρει στα λόγια, να ακολουθήσουν και αντίστοιχες πράξεις τώρα. Αναμένω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας ε, και παρά λοιπόν τις διστάμενες απόψεις ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα το ε, οποίο θα συμφενώσουμε όλοι. Έως τις 26 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας και τις 16 Μαΐου θα ψηφίσουμε ή μάλλον συγγνώμη θα ολοκληρώσουμε έτσι ώστε τον Ιούνιο να ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επί αυτής της ε, γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την παρουσίαση του προγράμματος Cultural and Creative Cities Monitor από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Σήμερα λοιπόν θα μας παρουσιάσει το κέντρο αυτό ένα νέο εργαλείο το οποίο δημιούργησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα. Ε, το εργαλείο αυτό έχει την ονομασία Cultural and Creative Cities Monitor. Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο ελέγχου και συγκριτικής αξιολόγησης επιδόσεων, benchmarking δηλαδή, το οποίο ε, έχει ενδιαφέρον ε, τόσο για τα μέλη της Επιτροπής ΚΟΥΤ όσο και για τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό της ε, ε, πολιτικής πολιτισμού για πολιτιστικά ζητήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ την κυρία Βαλατίνα Μοντάλτο και τον κύριο Στάιν Φερλάγεν από το γραφείο των Βρυξελών και να του δώσω κατευθείαν το λόγο. Δεν ξέρω βέβαια τι έχουν προβλέψει να κάνουν στο πλαίσιο των παρουσιάσεών του, αλλά θα έλεγα ο καθένα του έω ε, 7 ε, λεπτά και συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση. Σα καλωσορίζω και πάλι θερμά εδώ στη συνεδρίασή μα. Yeah. So, Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Μεγάλη τιμή και χαρά μου να είμαι εδώ. Η διαφάνεια κανονικά θα πρέπει να εμφανιστεί κάπου στην οθόνη. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι πιο δημιουργικές πόλεις στην Ευρώπη, οι πιο πολιτιστικές και τι αντίκτυπο έχει ο πολιτισμός στην οικονομία και την κοινωνία και το σημαντικότερο, πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο. Βλέποντας το έργο και τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, φαντάζομαι ότι έχετε συνηθίσει να αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Όταν θέλετε να συλλέξετε στοιχεία για να υποστηρίξετε ε, πολιτιστικές επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Στο κέντρο, κοινό κέντρο ερευνών, Τον Ιούλιο πέρσι ξεκινήσαμε ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης κατά χώρα που παρακολουθεί τις πόλεις, τις δημιουργικές και πολιτιστικές και συλλέγουμε ποιοτικά στοιχεία για να βοηθήσουμε τους αποφασίζοντες να δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ανέφερα. Πιο συγκεκριμένα το υποστήριξε ο Επίτροπος ο κ. Ναύρατσης το εργαλείο αυτό και έτσι η τοπική αυτοδίκηση έχει ένα εργαλείο οι πόλεις μπορούν να εκμεταλλευτούν το δημιουργικό τους δυναμικό. Θέλουμε να έχουμε καινοτόμε και ελκυστικές πόλεις και να καλύπτουν όλους και να είναι και ανθεκτικές. Ξεκινήσαμε κάνοντας ανάλυση. Εξετάσαμε επίσημα στατιστικά στοιχεία, κυρίως της Eurostat, και πειραματικά στοιχεία, όπως αποκαλούμε, από το διαδίκτυο κυρίως να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό και αξιόπιστα. Μια καινοτόμα πτυχή ήταν η προσπάθεια να δούμε και πέρα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και το TripAdvisor μας βοήθησε να συλλέξουμε στοιχεία. Φερρυπίν για τα μουσεία, για τα αξιοθέατα, για τις αίθουσες συναυλίων. Εντοπίσαμε μετά 168 πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις στην Ευρώπη σε 30 χώρες. Θέλαμε να εφαρμόσουμε ε, κριτήρια δικημενικά και διεθνώς συγκρίσιμα. Τι εντοπίσαμε 93 πόλεις που υπήρξαν ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Είχαν προεπιλεγεί για να γίνουν. 22 πόλεις που ανήκουν στο δίκτυο της UNESCO, δημιουργικών πόλεων, και 53 πόλεις οι οποίες φιλοξενούν τουλάχιστον δύο διεθνή πολιτιστικά φεστιβάλ. Το επόμενο, τι κάναμε. Ταξινομήσαμε τις πόλεις χρησιμοποιώντας 29 δείκτες. Επελέγησαν προσεκτικά οι δείκτες, ξεκινώντας από μια αρχική επιλογή 200 κριτηρίων. Η επιλογή βασίστηκε στη Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων και ανάγνωση διάφορων επιστημονικών συγγραμμάτων. Οι δείκτες μετά ομαδοποιήθηκαν σε νέα διαστάσεις που αφορούσαν τρεις βασικούς τομείς ε, που αφορούσαν τη ζωτικότητα των πόλεων. Πρώτα απ' όλα κοιτάξαμε ποια είναι η παρουσία διαφόρων ε, κτηρίων, ε, αίθουσε συναυλιών, μουσεία, θέατρα που μπορούσαν να οργανώσουν πολιτιστικέ εκδηλώσεις. Να δούμε σε ποιο βαθμό οι πόλει είναι, ζωτικής, είναι ζωντανέ όσον αφορά τα πολιτιστικά στοιχεία. Μετά, ε, απασχόληση απασχόλησης στο δημιουργικό τομέα, τον πολιτισμικό τομέα και ποια καινοτόμα προϊόντα έχουν δημιουργηθεί, νέα σχέδια, ε, διπλώματα τεχνίας, να δούμε πώ τελικά ο πολιτισμός συμβάλλει στην τοπική ε, οικονομία. Και μετά είδαμε με ποιο τρόπο οι πόλεις ε, υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Αν μπορούσαν, Φερρυπίν, να αναπτύξουν ανεκτό, ανεκτικό περιβάλλον προς την πολιτισμική ε, ποικιλομορφία. Τι βρήκαμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα προσπαθήσαμε να απεικονίσουμε την ιδεώδη δημιουργική πολιτιστική πόλη στην Ευρώπη, εντοπίζοντας τις επικεφαλής ε, πόλεις στις εννιά διαστάσεις. Τι βρήκαμε. Δεν υπάρχει μια μοναδική πόλη που να υπερέχει και σε νέα διαστάσεις. Η ιδεώδης όμως πόλης αποτελεί μείγμα οκτώ διαφορετικών πόλεων, κυρίως μεσαίου μεγέθους. Αυτή η πόλη θα έχει δημιουργικές θέσεις εργασίας όπως είναι στο Παρίσι, το ανθρώπινο κεφάλαιο, της Λεύεν, της Λουβέν, του Βελγίου και καινοτόμα προϊόντα της Ολλανδικής πόλης Eindhoven. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα είδαμε ότι το μέγεθος δεν είναι το μόνο που μετράει. Με άλλα λόγια, οι μεσαίου μεγέθους πόλεις θα πηγαίνουν αρκετά καλά εν συγκρίση με τις πιο μεγάλες. Κυρίως όσον αφορά τους δείκτες που δείχνουν τη ζωτικότητα την πολιτιστική. Τι είδαμε, ότι οι μεσαίου μεγέθους πόλεις ίσως να καλύπτουν περισσότερους, διότι παράγουν περισσότερο πολιτισμό ανακάτοικο. Ποιοι κερδίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε νέα διαστάσεις ε, που λάβαμε υπόψη. Είδαμε ότι έχουμε ένα κράμα διαφορών πόλεων. Κεφάλαια, ε, συγγνώμη, πρωτεύουσε και μη πρωτεύουσε. Παρίσι, Κοπενχάγη, Εδιμβούργο και Άιντχόβεν. Αυτές είναι οι πόλεις που είναι στις πρώτες θέσεις σε σχέση με άλλες πόλεις παρομοίου πληθυσμού. Παρίσι είναι πρώτο στην ομάδα πόλεων με περισσότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους θα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μία μοναδική κατηγοριοποίηση, αλλά πολλές βάσει ομάδων πόλων Φερρυπίν ε, με παρόμοιο πληθυσμό. Και στο διαδίκτυο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ομάδες πόλεων. Παραγωγή κατά κεφάλι κλπ. Κάναμε επιλογή, διότι το παρατηρητήριο δεν είναι ένα συγκριτικό εργαλείο, αλλά εργαλείο εκμάθησης μεταξύ ομοτήμων πόλεων. Κάθε πόλη έχει τα θετικά στοιχεία της και τις ιδιαιτερότητές της. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό. Η ανάλυση των στοιχείων τι επιβεβαιώνει, ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στην τοπική οικονομία. Από το 2009 μέχρι το 2013, Φερρυπίν, είδαμε ότι το ΑΕΠ ανακεφαλή αυξήθηκε πολύ ε, περισσότερο στις πόλεις που είναι πιο δημιουργικές. Το δείχνει ο δείκτης που συνοψίζει τη βαθμολόγηση ε, των 29 ε, δικτών. Οι πιο δημιουργικές πολιτισμικά πόλεις ήταν και πιο ανθεκτικές παρά την οικονομική κρίση. Αυτό διαπιστώσαμε. Όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέξαμε και αναλύσαμε είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στο εργαλείο, στο διαδίκτυο του παρατηρητηρίου μας αναβαθμίστηκε και έχει νέες λειτουργίες στο σελίδα μας. Τώρα μπορείτε εσείς να εισάγετε δικά σας στοιχεία εάν η πόλη σας δεν είναι στις 168 που έχουν επιλεγεί στην πρώτη έκδοση για να κάνετε σύγκριση με τις ε, πόλεις της πλατφόρμας ε, να δείτε ποια είναι τα θετικά και αρνητικά στοιχεία και τι μπορεί να βελτιωθεί. Άμα δείτε τι γίνεται σε άλλε αντίστοιχε πόλει, μπορείτε να δείτε και τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν οι πολιτικέ σα ε, όσον αφορά θέσει απασχόληση στο δημιουργικό τομέα και να δείτε πώ επηρεάζονται οι τελικοί βαθμοί. Το παρατηρητήριο αυτό ε, έχει γίνει καλά δεκτός όλη την Ευρώπη αρκετέ πόλει έχουν έρθει σε επαφή μαζί μα, όπω η Μπολόνια, η Μαδρίτη, η Βαλέτα, το η Πάλμα το, για να καταλάβουν πώς να χρησιμοποιήσουν καλύτερα το εργαλείο ή να εκφράσουν προθυμία να συμβάλλουν στη συλλογή στοιχείων για τις επόμενες εκδόσεις. Και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, στο Financial Times, την πρώτη σελίδα, εμφανιζόμαστε και σε άλλα ειδικά έντυπα και παρουσιάστηκε σε διάφορες ομιλίες και συναντήσεις όπως αυτή και σε εκδηλώσει πανεπιστήμια παρουσιάστηκε τα εργαλεία μας. Στο τέλος του έτους φέτος, θα ετοιμάσουμε και μία εφαρμογή του διαδικτύου, τόσο ώστε το παρατηρητήριό μας να πλησιάσει περισσότερο τους πολίτες. Στην εφαρμογή θα έχουμε τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να βοηθήσουμε τις αρχές των πόλεων να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες για θέματα πολιτισμού σε επίπεδο πόλης ή σε χαμηλότερο επίπεδο, να προωθηθεί ο πολιτισμός μέσω κυνηγιών θησαυρού πολιτιστικού περιεχομένου και να δώσουμε και οπτική εικόνα των βαθμών μέσω των εφαρμογών. Και το 2019 έχουμε τη δεύτερη έκδοση του εργαλείου αυτού, του παρατηρητηρίου, με επικαιροποιημένα στοιχεία και ίσως με ευρύτερο πεδίο κάλυψης. Τώρα προσπαθούμε να δούμε σε ποιο βαθμό το διαδίκτυο μας βοηθήσει να συλλέξουμε στοιχεία και όσον αφορά σε άτυπου, τους άτυπους χώρους πολιτισμού, όπως κοινοτήτων, για να συμπληρωθεί η εικόνα αντί να κινούμεθα μόνο στα μουσεία και στα θέατρα που έχουμε ήδη ε, στη βάση δεδομένων μας. Να διευρύνουμε τη βάση δεδομένων. Για άλλες πληροφορίες, πηγαίνετε στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στο διαδίκτυο, να το δείτε και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και η παρουσίαση του καινοτόμου αυτού εργαλείου του benchmark που βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων πόλων. Τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση. Να μην είμαστε τόσο επίσημοι, ε, δηλαδή να δώσω πρώτα το λόγο στους φεντονιστές για την ένας, α όχι δύο, τέλος πάντων. Όποιος ζητάει το λόγο θα παίρνει το λόγο, έτσι θα πάει. Η Ζαμπίνε Φερχάιεν πρώτη. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία. Έχω μια ερώτηση πολύ σύντομα. Είπατε ότι οι πόλεις ε, με τη μεγαλύτερη οικονομική ευημερία και που είναι ψηλά στην κατάταξη ό,τι αφορά ε, τον πολιτισμό είναι καλές πολύ εκεί. Δηλαδή συνδυάζονται αυτά τα δύο. Αυτό έχει να κάνει και με τη μεγαλύτερη οικονομική, ε, με τη χρηματοδότηση, δηλαδή η χρηματοδότηση ενισχύει την πολιτιστική πολυμορφία ή το αντίστροφο. Η κότα έκανε το αυγό κοτα κανει το αυγό την κότα. Θέλετε να απαντήσετε αμέσω, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ερώτηση. Είναι το αποτέλεσμα, χωρίς να πέσω λεπτομέρειες, οικονομετρικής αναλύσεως. Πάμε από την πολιτιστική πλευρά στα οικονομικά αποτελέσματα και όχι αντιστρόφως. Τι εξετάσαμε. Η Τα πολιτιστικά και ε, δημιουργικά στοιχεία πω επηρεάζουν το ΑΕΠ κατά κεφαλή. Η κίνηση είναι από πολιτισμό προς την οικονομική ανάπτυξη και όχι αντιστροφώ. Και εγώ έτσι κατάλαβα να είπατε ότι όσοι δήμοι ε, διακρίνονται για την πολιτιστική τους ε, ποικιλομορφία τα κατάφεραν ε, και καλύτερα στην οικονομική κρίση, γιατί είχαν επενδύσει, αν κατάλαβα καλά, όπως είπατε και εσείς, στα πολιτιστικά μόργανο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Έγινε αυτή η έρευνα εσωτερικά ή ανατέθηκε σε κάποιον. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. ηταν η Βασιζόμαστε εμείς επί της αξιοποίησεως της πολιτιστικής πολυμορφίας Πώς είναι η σχέση μεταξύ πολιτιστικής ποικιλομορφία και ορισμού ε, κριτηρίων για τους δείκτες όλη την Ευρώπη. Πρέπει να ευκρινιστεί αυτό. Τρίτον, σχέση με τα πανεπιστήμια. Όσον αφορά τι έρευνε που κάνατε, πόσο ευάρη είναι η παρουσία των πανεπιστημίων και των κέντρων των ερευνητικών στον εντοπισμό των διαφόρων στοιχείων. Είναι και θέμα του καθορισμού δικτών που καλύπτουν τον τομέα το δημιουργικό και τον πολιτιστικό μέσω δικτύου κέντρων αριστείας που αφορά και άλλα στοιχεία. Τελευταία πτυχή. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του έτους. Αν θέλουμε να κινηθούν και άλλες πόλεις, θα ήταν σωστό να ζητήσουμε μια επιτάχυνση αυτού Αλλιώ θα χάσουμε ένα χρόνο. είναι έτοιμη η εφαρμογή, το app, ε, πιο γρήγορα με λόγια. Απάντηση. Να απαντήσω Ιταλιστή ή σε άλλη γλώσσα. Όσον αφορά το ποιος έκανε την ε, έρευνα, εσωτερικά έγινε στο κοινό κέντρο έρευνας. Μία ομάδα τριμελής, τετραμελής το έκανε αυτό. Εσωτερικός. Δεν έγινε ανάθεση εξωτερικά. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά τις πόλεις, να μην ζητήσουμε συλλογή στοιχείων από τις πόλεις, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πηγές στοιχείων διαθεσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συλλογή στοιχείων έγινε σε κεντρικό επίπεδο από το Joint Research Center. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, το είπα και στον κατάλογο των δικτών. Αυτό ελήφθη υπόψη. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εκεί μετράμε την παρουσία των πτυχιούχων σε διάφορους τομείς, στον τομέα ανθρωπιστικών επιστημών, τέχνη, ανθρωπιστικές επιστήμες κλπ. Και μετρήσαμε και εντός των πόλων ποια είναι η παρουσία των πανεπιστημίων που έχουν κάποια προβολή σε εθνές επίπεδο. λαμβάνουμε υπόψη και τη θέση, την αριστεία των πανεπιστήμιων. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, είναι το θέμα. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε για να συμπεριλάβουμε δείγμα πόλεων το πιο αντιπροσωπευτικό που μπορούσαμε. Θέλαμε να συμπεριλάβουμε κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά και διαφορετικά. και ποια προγράμματα προωθήθηκαν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ε, πόλεων. Ε, ε, λοιπόν, συμπεριλάβαμε και το κριτήριο των πόλεων που έχουν τουλάχιστον δύο διεθνών φεστιβάλ. Και είδαμε ότι χρησιμοποιώντας τα εν λόγω κριτήρια που δεν εμπεριέχουν υποκειμενικότητα, καταλήξαμε σε ευρύτατο δείγμα πολλών πόλεων, επικύλων, ε, ΑΕΠ, κατά κεφαλή, ε, πληθυσμού κλπ. Έχουμε λοιπόν ευρύτατο δείγμα των πόλεων των δημιουργικών στην Ευρώπη. Η προσέγγιση μα ήταν τέτοια που θέλαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερου. Γι' αυτό δώσαμε τη δυνατότητα στι πόλει να βάλουν δικά του στοιχεία. Διότι θέλαμε να παίξουμε με κριτήρια αντικειμενικά. Αλλά οι δημιουργικέ και οι πολιτιστικές πόλεις περνάνε και το δείγμα αυτό που λάβαμε υπόψη. Για το app, για την εφαρμογή, ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του έτους η εφαρμογή αυτή για τα κινητά κλπ. Η app. Αν θέλουμε λοιπόν και οι πόλεις να δραστηριοποιηθούν και πιο γρήγορα, εάν δεν φτάσουν στο τέλος του έτους, ίσως θα ήταν καλύτερο. Ας πούμε τον Ιούνιο να είναι έτοιμο το app για να συμμετάσχουν οι πόλεις απάντηση. Αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τις πόλεις που είναι στο μόνιτορ τώρα. Η εξωτερική εταιρεία αναπτύσσει το app. Και αν άλλες πόλεις θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή αυτή σε τοπικό επίπεδο, αυτό θέλουμε, να μπορούν να συμμετάσχουν. Στείλαμε και ανακοίνωση στις επιλεγήσεις πόλεις για να τους πούμε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Και έτσι αν θέλουν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της εφαρμογής μπορούν να δηλώσουν και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής, της app. Ευχαριστώ. Πολύ απλό και σύντομο το ερώτημα που έχω και αφορά τα πολιτιστικά και δημιουργικά ζητήματα για τις πόλεις. Τη σημασία που έχουν οι πτυχές αυτές και κυρίως ό,τι αφορά την επιστημονική δημιουργικότητα, <clears throat> δηλαδή ε, δίκτυα ερευνητικών κέντρων, εξκαφές, ανασκαφές λοιπά. Τέτοιου είδους επιστημονικής δημιουργικότητας ε, έχει σημασία και σε ποιο βαθμό. Κοιτάξτε, η επιστήμη εξαρτάται από τον ορισμό και το εύρος αυτού. Όπως είπα, υπάρχει αυτή η διάσταση που λαμβάνουμε υπόψη, όπως η πτυχιούχη σε συγκεκριμένο τομέα και η θέση εργασίας. Όσο πίσω θέσεις έχουμε όσον αφορά τις τέχνες, ή δημιουργική, το δημιουργικό τομέα όπως είναι και η τεχνολογία ψηφιακή. Είχατε υπόψη έναν ορισμό όσον αφορά τις επιστήμες. Εμείς ακολουθήσαμε τεχνολογική δημιουργία υπόψη μας και ψηφιακή τεχνολογία. Ε, μιλάω για μουσεία επιστημών, φεστιβάλ, σχετικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να προβάλλουν αυτή την ανθρώπινη δημιουργικότητα, τεχνολογία, επιστήμη κτλ. Σίγουρα συμπεριλαμβάνεται. Δηλαδή, συμπεριλάβαμε τα μουσεία, δεν τα διθήσαμε μόνο μουσεία τέχνης Φερρυπίν. Όλα τα μουσεία αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Συμπεριλαμβάνονται. Εν αυτή τη έννοια, ναι, συμπεριλαμβάνονται. Ja, vielen, äh, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, για τις ερωτήσεις σας, για τις απαντήσεις που δόθηκαν. Νομίζω πως πρόκειται για ένα πολύ καλό project ε, και θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Αυτές οι δήμοι και οι κοινότητε ε, που δεν συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο monitoring, ε, πώς ενημερώνονται σχετικά με αυτό το project. Γίνεται δηλαδή τυχαία ή πρέπει να ε, δηλώσουν για παράδειγμα κάποια συμμετοχή ενεργά από τη δική τους πλευρά. Ε, προβαίνεται σε διαφήμιση ενεργά αυτού του εργαλείου προς τις ε, δήμους τους δήμους και τις κοινότητες. Και βέβαια ποια είναι η αντίδραση από την πλευρά τους, γιατί βέβαια πάντοτε τίθεται αυτό το ερώτημα, όταν δηλαδή κανείς υποβάλλεται σε μια συγκριτική αξιολόγηση, ε, και συγκρίνεται δηλαδή με άλλους ομοτήμους ε, είναι, είναι μια πρόκληση. Άρα λοιπόν ε, πώς αντιδρούν οι δημιουργικοί και πώς ενημερώνονται σε σχέση με την ύπαρξη αυτού του project, αυτού του εργαλείου. Κυρία Φαχάιν, θα ήθελα και εγώ να ζητήσω να μας πείτε αν υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος όλων των Δήμων που έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα. Yes, definitely. Σίγουρα, σίγουρα. Αν πάτε στο διαδίκτυο online, έχουμε και αντίγραφο της εκθέσεως εκεί στην είσοδο, αν θέλετε, έντυπα. Και θα βρείτε και τη λίστα των 168 πόλεων που επελέγησαν για την πρώτη έκδοση. Και online θα βρείτε λεπτομερείς εικόνες των 168 πόλεων, παρουσίασή τους, με ποιοτική περιγραφή και των βαθμών όσον αφορά τους 29 δείκτες. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα. Το κοινό κέντρο ερευνών προτείνει, να προτείνει κάτι σε πόλεις και να προωθήσει το προτινόμενο στο βαθμό του δυνατό. Οι απαντήσεις που παίρνουμε μας δείχνει η προθυμία που έχουν οι πόλεις να συμμετάσχουν περισσότερο στην προσπάθεια και να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιείται το εργαλείο. Κατά κάποιο τρόπο ξεκινάμε δημιουργία δυναμικού μέσω μιας διαδικασίας, διότι έρχονται οι πόλεις, μας ζητούν να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία χρησιμοποιούν ε, διαφορετικά το εργαλείο. Καμιά φορά το χρησιμοποιούν για να βρούνε παρόμοιες πόλεις που τα πηγαίνουν καλύτερα ή πώς μπορούν να δείξουν ότι τα πάνε καλά κάποιες πόλεις ή κάπου να εντοπίσουν πόλεις που θα μπορούσαν καλοί εταίροι σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήταν άλλη μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που συλλέξαμε. Άρα για την ώρα ε, διαδίδεται το είδηση ταχαίως και αν δεν σε επαφή μαζί μας του τους λέμε να, έρθουν σε επαφή μαζί μας ή να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να βάλουν τα στοιχεία τους. Και έχουμε ενδιαφέρον αίτημα από την περιοχή Εμίλια Ρωμάνια που θέλει να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο σε όλες τις πόλεις της περιοχής και να χρησιμοποιήσουν τα δικά του στοιχεία και να δουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα της χρήση του μοντέλου για τις πόλεις της περιφέρειας αυτής, Εμίλια Ρωμάνια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ Πέτρα, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είμαι μέλος της διακοινοβουλευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου για τη Δημιουργική Βιομηχανία. Για μία δεκαετία περίπου συζητώ με του εκπροσώπου του τομέα τα θέματα αυτά, πώς μπορεί η δημιουργικός τομέας να οδηγήσει οικονομική ανάπτυξη, κάλυψη του κοινωνικού ιστού και βελτίωση της καταστάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Τι είδαμε στις τελευταίες εκλογές κυρίως στις πόλεις, είναι πιο ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Στην Ήπεθρο και σε μειονεκτούσες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα όταν αναφέρεστε το ρόλο των πόλεων. Τι γίνεται με τον κόσμο που δεν ε, ζει στις Μητροπόλεις και στις υπέροχες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά ζουν στην Ήπεθρο, σε μειονεκτούσες περιοχές. Το εισηγητής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης Είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό και θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται οι νέοι σε μειονεκτούσες περιοχές. Εάν δεν πλησιάσουμε την Ήπεθρο, έχουμε πολιτικής φύσεως πρόβλημα. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη σε κάποιο βαθμό, με κάποιο τρόπο. Απάντηση. Η απάντηση είναι όχι. Για απλούστατο λόγο. Εστιαστήκαμε επί των πόλεων. Ξέρετε τι ρόλο αποκτούν οι πόλεις τελευταίες δεκαετίες. Γι' αυτό όχι γιατί απορρίπτουμε την περιφέρεια ή την Ήπεθρο, αλλά θέλαμε από κάπου να ξεκινήσουμε με ένα μοντέλο που να μπορεί να εφαρμοστεί εκεί που υπάρχουν οι πληροφορίες. Στις πόλεις έχουμε θέσιμα στοιχεία. Για την Ήπεθρο είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν θεσμική άποψη. Είναι κάτι που θα πρέπει να καλυφθεί η στην αρχή ήταν δύσκολο να το κάνουμε αυτό, να καλύψουμε και την ύπεθρο, αλλά δεν απορρίπτουμε καθόλου αυτή την κάλυψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και την παρουσίαση αυτού του project. Ε, νομίζω ε, πως όλοι μας εδώ σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ε, ελπίζοντας πως θα συμμετάσχουν ακόμα περισσότερες πόλεις στο μέλλον, σε αυτό το project, έτσι ώστε βέβαια να ξεκινήσει ένας, ε, μια ανταλλαγή απόψεων, ένα διάλογο μεταξύ του και όχι απλά ένα ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τι επιδόσει του. Ε, θα μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο οι πόλεις να δουν ε, τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα, τι μπορούν να βελτιώσουν οι ίδιε ή που οι ίδιε καταφέρνουν κάτι καλύτερα σε σύγκριση με του υπόλοιπου. Σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σα σήμερα εδώ και σα εύχομαι κάθε επιτυχία στι μελλοντικέ εργασίε. Τώρα, Συνεχίζουμε και μένουμε στα του πολιτισμού. Περνάμε δηλαδή σε μία συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ πρωτοβουλίε στην πολιτισμική και δημιουργική οικονομία. Και εδώ καλωσορίζω θερμά τον κύριο Μάρτιν Κιάν, ο οποίο ήρθε εδώ από τη Βουδαπέστη και ο οποίο είναι ε, προσωρινό διευθυντή του EIT, αυτού δηλαδή του Ινστιτούτου. Θα μα ενημερώσει για τι δραστηριότητες του EIT, αλλά και τις ε, προσπάθειες ε, που κάνει, τη φιλοδοξία του να δημιουργήσει στο μέλλον μία κοινότητα καινοτομία για, για την πολιτισμική και την δημιουργική βιομηχανία. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κιάν για 5 έως 7 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την για την πρόσκληση να στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έρθουμε να παρουσιάσουμε τη θέση μας σαν Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομή Τεχνολογία και να παρουσιάσουμε μελλοντικέ στρατηγικέ για πολιτιστικό, πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Να σα δώσω μια επισκόπηση, να σα παρουσιάσω επισκόπηση. Τι είναι το EIT, ίσω να μην το ξέρετε τόσο καλά, τι έχει πετύχει, και μετά να δούμε ποια είναι η μελλοντική μας στρατηγική. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικότατος, διότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ξεκινώντας λοιπόν, από την αρχή, να σας πω λίγα λόγια για το υπόβαθρο. Γιατί δημιουργήθηκε το EIT, δημιουργήθηκε διότι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστερεί όσον αφορά την καινοτομία. Um, λοιπόν, η Ευρώπη πάει πολύ καλά στην έρευνα Είδαμε ένα άριστο παράδειγμα του ερευνητικού εργαλείου. Δεν τα πάει τόσο καλά η Ευρώπη όσον αφορά τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, σχέση με περιοχέ του κόσμου, κυρίω με τη ΣΥΠΑ, την Ασία και το Ισραήλ, αν συγκρίνουμε. Το EIT, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, δημιουργήθηκε το 2008 με αυτό το υπόβαθρο που περιέγραψα. Προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Άριστη έρευνα αρίστων πανεπιστημίων στην Ευρώπη, χωρί πολλή καινοτομία. Θα δημιουργήσει συμπράξει πανευρωπαϊκές που προωθούν στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και εταιριών. Είναι κοινότητε γνώση και καινοτομία όπω τι αποκαλούμε. Θέλουμε να είναι πιο ασχολούνται με επιχειρηματικά οι σπουδαστέ και νεοφύσει εταιρείε να αυξάνονται, να επιτυχαίνουν τα, τις ανακαλύψεις του εργαστηρίου να τις διαθέτουμε στην αγορά. Αυτή είναι η εντολή βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το ΙΕΤ. E Δέκα χρόνια μετά το πετύχαμε, δημιουργήσαμε μια πολύ ευρία κοινότητα καινοτομίας και έρευνας, έχουν πάνω από χίλιους εταίρες, εταίρους, οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις, νεοφύης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, τη βιομηχανία και έχουμε και κόμβους, πάνω από 40 κόμβους καινοτομία στην Ευρώπη. Σε επιχειρησιακό επίπεδο έχουμε έξι κοινότητες καινοτομία που ασχολούνται με προβλήματα για την κοινωνία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το EIT. Ασχολούμαστε με την ψηφιοποίηση στην αλλαγή του κλίματος, υγεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και πρώτες ύλες. Αυτές είναι οι προκλήσεις για την κοινωνία και θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο νέες κοινότητες καινοτομία για την αστική κινητικότητα και την μεταποίηση και την παραγωγή. Είναι θέματα στα οποία η καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά να αφελήσουν την Ευρώπη. Ισχυρότατο οικοσύστημα καινοτομία είναι αυτό που δημιουργήθηκε και που δίνει επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία. Δεν το λέμε απλώς. Έχουμε και στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό επιτυγχάνεται, διότι πέρσι δύο μελέτες ολοκληρώθηκαν όσον αφορά το ΙΕΤ e από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μια μελέτη με τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και η δεύτερη μελέτη, η μελέτη αντικτύπου όσον αφορά τα συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα που έχει πετύχει το EIT και η μελέτη καταδεικνύει ότι όχι μόνο αυτές οι κοινότητες καινοτομία δημιουργήθηκαν και υποστήριξαν πάνω από 100 επιχειρήσεις και πάνω από 6.000 θέσεις ε, απασχόλησης αλλά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ προσήλκησαν σε επενδύσεις εταιρείε και στις νεοφυείς ε, επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν και στην αγορά ε, διαθέσαμε 400 καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το EIT δίνει αποτελέσματα, λειτουργεί και το EIT ε, δίνει λύσεις όσον αφορά τα προβλήματα τα κοινωνικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Ένα παράδειγμα είναι οι διάφορες τεχνολογίες για αποθήκευση ενέργειας και ε, μπαταριών που υποστηρίχθηκε από το EIT, ε είναι ένα καλό παράδειγμα. Από μια μικρή πόλη της Εστονίας ξεκίνησε. Από το Πανεπιστήμιο του ΤΑΤΟΥ έγινε έρευνα από τη δεκαετία του 90 για την αποθήκευση της ενέργειας, ε, πυκνοτές μεγάλης χωρητικότητας, αλλά αφού εντάχθη ναι, η πόλη αυτή στην ε, κοινότητα του ΑΕΤ και σε επαφή με το όλο οικοσύστημά μας της καινοτομίας, το μικρό ερευνητικό πρόγραμμα έγινε τυχέστατο πρόγραμμα και έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και έχει 100 άτομα προσωπικό και δημιουργεί συσκευές αποθήκευσης ενέργειας που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και χρησιμοποιείται το προϊόν κυρίως στον τομέα της κινητικότητα ένα παράδειγμα επιτυχίας. Πώς ε, έρευνα μέσω διασυνδέσεων, μέσω της επαφή με την κοινωνία ε, μπορεί να είναι επιτυχής. Και βλέπετε από τον πρόεδρο της εταιρείας ότι αναφέρει ότι βοήθησε η IT ε, και υποστηρίχθηκε η εταιρεία από το e IT για να πετύχει η εταιρεία. Είναι αυτές οι τεχνολογίες σκελετού όπως αποκαλούμε, δημιουργούν τη ραχοκοκαλιά της προσέγγισης. Και έχει και μια διάσταση εκπαιδευτική ο μας. Έχουμε πρόγραμμα για την εκπαίδευση όσον αφορά τον, την επιχειρηματικότητα. Μπορεί να σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Προσπαθώ να συνδυάσουμε αριστεία, τα πτυχία, τους πτυχιούχους, τους αρίστους ε, των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι πτυχιούχοι λοιπόν έχουν την τεχνογνωσία, μπορούν να είναι επιστήμονες υπολογιστών, μηχανικοί, Πρέπει όμω να καταλαβαίνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα. Εκεί του βοηθούμε. Να είναι οι καινοτόμοι του αύριο. Να είναι εκείνοι που θα μπορούν ε, αύριο να δημιουργούν καινοτομίε, καινοτόμα προϊόντα που θα λύνουν τα διάφορα προβλήματα τα κοινωνικά. Τα προγράμματα που έχουμε και εφαρμόσει σε πανεπιστημιακό επίπεδο αξιολογούνται, θεωρούνται μοναδικά, εστιάζονται επί δεξιοτήτων, επί δημιουργικότητα και καινοτομία. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν μια ισχυρότατη διάσταση κινητικότητα ο, ο σπουδαστή πρέπει να πάει τουλάχιστον σε δύο χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να πάρει ένα διπλό πτυχίο, αν θέλετε, και ε, μια, ένα πιστοποιητικό του EIT που, έχει, που δείχνει ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα της μιλικότητας και της καινοτομίας. Επίσης, όλο και περισσότερο τονίζεται η ψηφιακή εκπαίδευση. Το EIT ε, Digital είναι μία από τις καινοτόμους κοινότητες με προγράμματα Έχουμε ακαδημία ψηφιακή του EIT που αναμειγνύει την εκπαίδευση στο διαδίκτυο με την κλασική εκπαίδευση στην τάξη και με τη διάσταση επιχειρηματικότητα. Συνδυάζει όλα αυτά. Πρόσφατα το EIT έχει προωθήσει και άλλε μορφέ εκπαίδευση για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Εργαζόμαστε με 12χρονες μέχρι 18χρονες για να προωθήσουμε ψηφιακές δεξιότητες, να τους δώσουμε παραδείγματα επιτυχούς θηλυκής επιχειρηματικότητας και να τις ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν σε καινοτόμους τομείς και σε διάφορα προγράμματα πανεπιστημιακά. Αυτό κάνουμε. Θέλω να δω τι θα κάνουμε στο μέλλον. Διότι τώρα το EIT ετοιμάζει στρατηγική για την περίοδο μετά το 2021 και έχει υποβάλει την πολιτική το Δεκέμβριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη νέα στρατηγική λοιπόν έχουμε τέσσερις στόχους που έχουμε θέσει. Οι τέσσερις στόχοι βασίζονται επί της αρνής του βάσεως που δημιούργησε το EIT. Θέλουμε να εδραστούμε επί των χρησιμοτάτων αυτών εργαλείων και μοντέλων των προτύπων που έχουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα οικοσυστήματα ε, καινοτομία που δημιουργήσαμε, να τα καταστήσουμε ισχυρότερα και να καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Έχουμε ήδη μια καλή βάση γι' αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και τα οχτώ προβλήματα που έχουμε, αλλά και τους άλλους τομείς. Πολιτισμός και δημιουργικός τομέας και δημιουργική βιομηχανία, θα αναφερθώ σε αυτό σε λίγο, και να συνεχίσουμε την εκπαίδευση στον επιχειρηματικό τομέα, να έχουμε επιτυχή προγράμματα και να καλύπτουμε και κάτι παραπάνω από τα πανεπιστήμια στα οποία εστιαστήκαμε και έχουμε, όσο περισσότερο έχουμε επιτυχείς καινοτομίες, τόσο θέλουμε να τις διαδώσουμε για να ωφελείται όλη η Ευρώπη από τις επιτυχείς καινοτομίες και να υπάρξουν και συνέργειες με άλλα προγράμματα. Λοιπόν, σαν τμήμα της στρατηγικής, μία από τις νέες καινοτόμες κοινότητες που δημιουργήσαμε είναι για το πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και αυτό επηρεάζει πολύ τον τομέα που σας ενδιαφέρει, τον τομέα με τον οποίο ασχολείται η Επιτροπή Κουλτ Θέλω να παρουσιάσω κροθυγό τον τομέα αυτό και θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι απόψει σα και να ακούσω τυχόν ερωτήσει σα, Τι προτείνουμε. Μια κοινότητα καινοτομία του ετή για το δημιουργικό και ε, πολιτιστικό τομέα να είναι ένα τμήμα συνολική στρατηγική. Στην ανάλυση που κάνουμε, μια τέτοια κοινότητα καινοτομία θα μπορούσε να ταιριάζει πάρα πολύ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι δημιουργικότητα είναι στο επίκεντρο του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και πώς η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα η Ευρώπη έχει εξαιρετικά ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά και πολύ ισχυρό πολιτισμικό περιεχόμενο. Δεν είναι πολύ καλή Ευρώπη να το μεταφράζει αυτό σε καινοτομία και καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες που χρειάζονται οι πολίτες και μπορούν να ωφελήσουν τους πολίτες. Προφανώς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση στον τομέα αυτό. Εν γέννη όμως βλέπουμε ότι οι επιδόσεις της Ευρώπης δεν είναι ιδεώδεις. Άρα υπάρχει τεράστια δυνατότητα να καλύψουμε κενά στον τομέα και το μοντέλο του EIT στην πανευρωπαϊκή κοινότητα καινοτομία θα μπορούσε να βοηθήσει να ελευθερώσουμε το δημιουργικό που υπάρχει, το δημιουργική δυναμικότητα. Μπορεί να είναι πιο ορατή Ευρώπη στο παγκόσμιο προσκήνιο και να γίνει πρέσβης αξιών μέσω του πολιτισμού και της πολιτισμικής της κληρονομιάς ε, προβάλλοντάς τα όλα αυτά. Τι μπορεί να περιμένει κανείς από μια κοινότητα καινοτομία στο πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα, αν προχωρήσουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό που πολύ συχνά υπάρχει στον τομέα αυτό και να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα, για τους ε, εκπαιδευτές, τους φοιτητές, τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να δημιουργηθούν νέα κυβερνητικά μοντέλα συμπράξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα και κυρίω να συμμετέχουν οι πολίτε σε όλη την Ευρώπη στο πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα και σχετικέ δραστηριότητε. Μπορεί να δημιουργηθεί πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο, δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, ανάπτυξη, νέε επιχειρηματίε, νέε επιχειρήσει, νέε τεχνολογίε να αναπτυχθούν στον τομέα και τι προσφέρουμε είναι συστημικό ή μακροπρόθεσμο, διότι μια κοινωνία καινοτομία για 7 με 15 χρόνια αφορά 400 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα επιτρέπει να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα και μεταμόρφωση. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Λοιπόν, προσφέρουμε επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση επιχειρηματικότητα, επιτάχυνση της αναπτύξης των νεοφιών επιχειρήσεων και παραγωγή καινοτομία. Και όλα αυτά θα μεταφραστούν σε νέα προϊόντα, υπηρεσίε και αγορέ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να αναπτυχθεί οικονομικά, αλλά να αναπτυχθούν οι χώρε μαζί μέσω τη τη πολιτισμική κληρονομιά. Είναι ένα θετικό θεματολόγιο που, κάτι που χρειάζεται πολύ η Ευρώπη. Και θα ήθελα να ακούσω ποιε είναι οι απόψει σα, τι ιδέε έχετε και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει. Σα ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την παρουσίαση των όσων ε, σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον. Δύο συναδελφοί έχουν ζητήσει το λόγο. Καταρχήν η Χέλικα Τρίπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ε, θέσω κάποια ερωτήματα. Όταν ανέλαβα ε, το 2004 ως Ευρωβουλευτής είχαμε θέσει ως στόχο ως το 2010 να είμαστε η μεγαλύτερη κοινωνία βασισμένη στη γνώση και αποτύχαμε σε σχέση με αυτό το στόχο ε, και είμαστε στο 2018 και παραμένουμε ε, ως ε, δεν είμαστε η μεγαλύτερη κοινότητα βασισμένη στη γνώση. Και θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι λήψει. Μα είπατε ότι έχουμε πολλέ ε, κοινοτομίε, αλλά δεν μπορούμε να τι φέρουμε στην αγορά, γιατί υπάρχουν μονοπόλια, υπάρχουν στρεβλώσει του ανταγωνισμού και ούτω καθεξή. Και υπάρχουν και κάποιε ε, υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα από την πλευρά μας ως Ευρωπαίοι. Ε, θα ήθελα να μου πείτε όμως ε, ποιοι είναι οι λόγοι που σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί μας είπατε αυτό ότι δηλαδή θα υπάρξει πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος, θα υπάρξουν τέτοιου είδους κοινότητες καινοτομία και ούτω καθεξής. Ναι, εντάξει, είναι θετικά όλα αυτά. Μας είπατε ότι θέλετε να έχουμε public-private partnerships, εταιρικέ σχέσει δηλαδή δημοσίου ιδιωτικού τομέα και μα είπατε ότι θα προσπαθήσετε να ε, ευαισθητοποιήσετε περισσότερο του πολίτε μα. Ε. Μα όλα αυτά τα κάνουμε ήδη. Ε, γιατί λοιπόν θα υπάρξει περισσότερος αντίκτυπος αυτής της πολιτικής. Ε, γιατί να σας πιστέψω δηλαδή σε αυτά που λέτε τώρα όταν πριν από 10 χρόνια απέτυχαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Λιμπάτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κέρνα για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017 ανακοίνωσε ότι το EIT, αυτό το Ινστιτούτο, θα διευρύνει τον, το πεδίο της αρμοδιότητάς του, προκειμένου δηλαδή να καλύπτει και τελειόφυτους ε, και κατόχους διδακτορικών ε, τίτλων προκειμένου να υποστηρίζει τα project τους. Άρα συμβαίνει αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεύτερο ερώτημα. Η κυρία Τρούπελ ε, το ανέφερε ήδη ότι υπάρχει ένας πραγματικός κατακαιρματισμός αυτής της, αυτού του τομέα, δηλαδή εδαφικός κατακαιρματισμός. Οπότε τι θέλετε να κάνετε για να αντιμετωπιστεί αυτό. Και τρίτο ερώτημα, ναι, είναι ε, θετικό αυτό που αναφέρατε, ότι δηλαδή θα πρέπει η γνώση να γίνεται αντιληπτή και να αντιμετωπίζεται ως ε, πολιτισμικό αγαθό. Αλλά πώς ακριβώς αυτό θα το κάνετε στην πράξη, πώς δηλαδή προωθείτε την επιχειρηματικότητα σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέρν για να απαντήσει σε αυτά τα δύο ερωτήματα που δεν ήταν σε ε, καμία περίπτωση ιδιαίτερα εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα για να συσχετίσουμε το έργο του EIT με την γενική κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Ε, είναι λίγο υπερβολικό, είναι κάπω παρατραβηγμένο. Δεν μπορεί μόνο το, Ινστιτούτο να υπερκεράσει το χάσμα που υπάρχει, την έλλειψη σε επαρκή έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη. Την ε, συμβολή του σίγουρα ε, μπορεί να την προσφέρει. Είπα ότι έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, ότι έχουμε προσφέρει Είμαστε όμως ένα μικρό κομμάτι του προγράμματος Horizon 2020, 4% συγκεκριμένα και ο στόχο σίγουρα είναι να βοηθήσουμε την Ευρώπη να προχωρήσει στον τομέα τη έρευνα και καινοτομία. Αλλά το EIT από μόνο του δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα ε, αν δεν μπορεί και το ορίζον 2020. Κάποια πρόοδο, κάποια μετακίνηση βλέπουμε. Αλλά το δίλημα που είπατε και το οποίο έχει ε, εντοπιστεί ήδη εδώ και 10 χρόνια εξακολουθεί να ισχύει. Δεν έχουμε καινοτόμη, επαρκή ε, καινοτομία και σχετικές δυνατότητες. Είμαστε πίσω. Τι άλλα εμπόδια, λέει η κυρία Τρόπλη, σας είπα. πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, να εστιάσουν περισσότερες προσπάθειες και είχατε δίκιο ότι στο ψηφιακό τομέα η Ευρώπη έχει μείνει πίσω κατά πάσα πιθανότητα. Άλλοι ε, στον κόσμο έχουν τα ε, έχουν την ηγετική θέση. Υπάρχουν όμως νέοι τομείς και οι πολιτιστικές ε, βιομηχανίες ε, είναι ένα τομέα, αλλά έχουμε την υγεία, τα τρόφιμα, την ενέργεια, το περιβάλλον, το κλίμα. Εκεί θα μπορούσε να πάρει ε, ηγετική θέση η Ευρώπη και να γίνει ηγέτης και πρωταγωνιστής σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Αυτό προτείνουμε και προτείνουμε να αναβαθμίσει τι προσπαθίε τη Ευρώπη, γιατί χρειάζονται περισσότερα. Θέλουμε μεγαλύτερε επιτυχίε, περισσότερη καινοτομία και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφο. Ό,τι αφορά στην έκθεση του 2014 δύο θέματα έφυγε. Πρώτον ότι το EIT ε δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να καταδείξει ότι είχε αποτελέσματα και μπορεί να επηρεάσει και υπήρχε και κάποια πολυπλοκότητα στις ε, δραστηριότητες μας. Κάναμε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο προβλήματα. Ήταν μια νέα πρωτοβουλία το EIT, άρα χρειάστηκε να περάσει κάποιο διάστημα, να κάνουμε τις σχετικές διορθώσεις. Τώρα βλέπουμε τον αντίκτυπο, βλέπουμε τα τα αποτελέσματα και αυτό το επικύρωσαν οι δύο μελέτες πέρυσι. Επίσης καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες για να είμαστε απλοί στις διαδικασίες μας. Έχουμε χίλιους εταίρους ε, και έξι κοινότητε καινοτομία. Φαντάζεστε ότι όλα αυτά σημαίνουν κάποια πολυπλοκότητα. Θέλουμε όμω να είμαστε αποτελεσματικοί και καινοτόμοι και αυτό θα το πετύχουμε αν είμαστε απλοί στον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τις κοινότητε αυτές και νομίζω ότι καταφέραμε να περιορίσουμε σημαντικά την πολυπλοκότητα και τα αποτελέσματα τα μπορείτε να τα δείτε. Ένα άλλο ερώτημα ήταν ποιε είναι οι διαφορές στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ ό,τι αφορά την δυνατότητα καινοτομία στην Ευρώπη. Ναι, πράγματι το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Υπάρχουν οι κόμβοι καινοτομία στο Βερολίνο, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Αυτή είναι η ηγέτης καινοτομία αλλά σε χώρες όπως Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία χρειάζεται κάτι αντίστοιχο, να υπάρξει ενίσχυση της ε, συνεργασίας ε, ακαδημαϊκών, ερευνητών. Ε, έτσι, το 2014 ξεκίνησε αυτό το σχήμα καινοτομία το Innovation Scheme και έχουν ενταχθεί και χώρες τώρα που δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα. Και το ποσό που πηγαίνει στις 13 χώρες είναι το διπλό από ότι ο μέσος όρος ε, του ορίζοντα 2020. Κάνουμε προσπάθειες λοιπόν να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να δώσουμε δυνατότητα και ατομία σε όλη την Ευρώπη, γιατί το EIT ε είναι ένα Ινστιτούτο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σβέρ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει το Ινστιτούτο σας. Και αυτό που είπατε, αυτό ακριβώς χρειάζεται ισχυρά κέντρα καινοτομία, κόμβη, σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ε, αν θέλετε, ένας ανταγωνισμός στον τομέα της καινοτομία και εμείς είμαστε χαμένοι από ό,τι φαίνεται απέναντι στην Ασία, για παράδειγμα, ή και άλλα κράτη. Η Κίνα επίσης κερδίζει έδαφος σε ό,τι αφορά την καινοτομία και αλλα κρατη η κινα επιση κερδιζει εδαφος σε οτι αφορα την καινοτομια και παραπανω και η Ευρώπη. Είναι η γυραιά κυρία που δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα. Έτσι παρουσιάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι σε ό,τι αφορά δημιουργία υποδομών ή χάραξη πολιτικών, αλλά η καινοτομία θέλουμε να αποτελεί έναν τρόπο ζωής ουσιαστικά. Ο Μαξ Φέμπερ έλεγε να υπάρχει αυτή η καινοτομία το γίγνεσθε. Έτσι πρέπει. να το εντάξουμε στην όλη τη λογική της δουλειάς μας. Και αυτό να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε χάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει ακόμη και τα μικρά παιδιά να μπορούν να είναι καινοτόμα για να προχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόργανο. <clears throat> Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι στην παρέμβασή σας εντοπίζουμε πολιτισμό, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Τέσσερις λέξεις που επισημαίνουμε. Και σε κάποιο βαθμό επιμένετε στην εισαγωγή σας επί της δημιουργικότητας. Θεωρείτε ότι ίσως η καινοτομία, πώς να το πω, η καινοτομία ήταν ένα είδος, πώς να το πω, συνέπειας. Μετά όμως η ομιλία αναφέρεται στην καινοτομία του προϊόντος και την τεχνολογική καινοτομία, το λέω αυτό. Δημιουργείται αυθόρμητα το ερώτημα. Εκτίθεται το Ευρωκοινοβούλιο σαφέστατα μέσω ενός ψηφίσματος για τα θέματα της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. Και είπαμε σαφέστατα κάποια πράγματα στο ψήφισμα. Ζήτησε να υπάρχει στρατηγική επιλογή που θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το ΕΦΣΥ αμυστατικών επενδύσεων και να κάνει κάποια πράγματα μεγάλα ε, τα ποσά που αναφέρονται. Δεν αληθεύει ότι όσον αφορά τη δημιουργική βιομηχανία και τον πολιτισμό έχουμε στη δεύτερη θέση σε σχέση με άλλους. Ερώτημα λοιπόν που τίθεται το Ινστιτούτο λοιπόν όσον αφορά αυτά τα θέματα και σε σχέση με το αίτημα χρηματοδοτήσεως. Ασχοληθήκαμε με το ΕΦΣΙ. Στο ΕΦΣΙ 2 ζητούμε να γίνουν κάποια πράγματα να βρεθούν κάποιες λύσεις προθυμένες που αφορούν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάνουν στατικές επιλογές άλλες χώρες διαφορετικές. Για να θα πρέπει να αλλάξουν παραγωγικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταγωνιστούμε τι άλλε χώρε Στο τέλο, με 20 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό πλαίσιο. Τι προτίθεστε να κάνετε το να επιμείνουμε επί κάποιων θεμάτων ότι πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει να κάνουμε πράγματα, αυτό δεν είναι αρμοδιάτητα της πολιτικής ούτε εκείνου που χειρίζεται ένα Ινστιτούτο. Για να γίνει κάτι χρειαζόμαστε το ένα, το άλλο και το άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που συσχετίζει ε, κάποια στοιχεία. Υπάρχουν κέντρα έρευνας που εργάζονται, λειτουργούν, παράγουν και μια άλλη πτυχή υπάρχει και επιμένω από αυτού. Μην λησμονούμε ότι η καινοτομία είναι η καινοτομία του προϊόντος και έχουμε αριστεία στην Ευρώπη που αναγνωρίζεται. Δεν το λέω αυτό για να αμυνθώ. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Μήπως κινδυνεύουμε να κάνουμε, να καλύπτουμε έναν πολύ, να καλύπτεται ένα πολύ περιορισμένο κύκλο. Συγγνώμη την ειλικρίνη, αλλά πρέπει να τα πω αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα από τη δική μου πλευρά. υπάρχουν μια σειρά από φήμες ε, που κυκλοφορούν σε ό,τι αφορά το μέλλον των ε, διαφορών προγραμμάτων ε, και μία από αυτές τις φήμες που άκουσα εγώ τουλάχιστον είναι ότι ο τομέας της, του πολιτισμού και της καινοτομίας δεν θα υφίσταται ως τέτοιο στο νέο πρόγραμμα Horizon 2020. Άρα σας θέτω το εξής ερώτημα. πώς συμβιβάσετε κάτι τέτοιο με τον ε, προσανατολισμό σας για το μέλλον, ε, δηλαδή να ασχοληθείτε περισσότερο από την πλευρά του Ινστιτούτου σας με το τομέα της δημιουργικότητας και της ε, κοινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι χρηματοδοτήσετε από το Horizon 2020. Και σας ρωτώ πιο συγκεκριμένα, γνωρίζετε αυτή τη φήμη, την ακούσατε και ενδεχομένως θα την γνωρίζετε γιατί προέκυψε. Πάντως θα έχει αποφασιστική σημασία αυτό, δηλαδή αν θέλουμε περισσότερο να ασχοληθούμε με τα ζητήματα της κοινοτομίας, να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο Horizon γι' αυτό. Αλλιώς θα βρισκόμαστε σε μια αντίφαση. Ο λόγος του κύριο Τιά. Ε, ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσβέρη για τα ερωτήματα που έθεσε και τις παρατηρήσεις του. Ουσιαστικά συμφωνώ μαζί του, περιέγραψε πολύ καλά το τι προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια επιχειρηματική κουλτούρα εδώ στην Ένωση ε, και πράγματι συνεργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό φοιτητέ με νέου και startups, νεοφυεί επιχειρήσει και βλέπουμε ένα τεράστιο ενθουσιασμό να ε, πράγματι αναβιώσει περισσότερη επιχειρηματικότητα και να υπάρξουν περισσότερε ε, ιδέε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν δεν δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία, το απαραίτητο οικοσύστημα σε αυτού του φοιτητέ, τότε υπάρχει ο κίνδυνο να μην παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μεταβούν κάπου αλλού, για παράδειγμα στο Silicon Valley, για να υλοποιήσουν αυτέ τι ιδέε του. Αυτό είναι ο κίνδυνο και προσπαθούμε λοιπόν να διαθέσουμε αυτό το οικοσύστημα ε, ε, δημιουργικότητας και νοτομίας αυτούς του νέους προκειμένου να παραμείνουν εδώ και να ε, μεταφράσουν στην πράξη αυτές τις ιδέες τους. Και το κάνουμε αυτό και με την ανάπτυξη των καταλήγων μορφωτικών προγραμμάτων. Και τώρα, τι κάνουμε συγκεκριμένα εδώ. Σε ό,τι αφορά την κοινότητα καινοτομίας πρέπει δηλαδή ο, η διάρκεια τη είναι 7 έως 15 έτη. Από εκεί και μετά θα πρέπει από μόνη της να λειτουργεί χωρίς υποστήριξη από την πλευρά της Δηλαδή ουσιαστικά η υποστήριξή μας αξιοποιείται ως καταλήτης για να προσελκυθούν περισσότερες επενδύσεις και περισσότερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από τα ερευνατικά κέντρα, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτά τα προγράμματα, να δημιουργηθεί αυτή η επιχειρηματική κουλτούρα στην Ευρώπη, προκειμένου ε, οι άνθρωποι, όπως σε αυτό το τομέα της ε, δημιουργικότητας και της να επιθυμούν να ε, δραστηριοποιηθούν ε, επιχειρηματικά. Δημιουργούμε λοιπόν τέτοιου είδου ε, τεχνολογίε ε, σκελετού, δηλαδή τεχνολογίε βάση για κάτι περαιτέρω. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε δηλαδή success stories όπου προωθούμε την ανάπτυξη και δημιουργούμε θέσει εργασία. Δημιουργούμε δηλαδή αυτά τα πλαίσια προκειμένου οι επιχειρήσει, ο ερευνητικό τομέα να συνεργάζονται μεταξύ του με τι νεοφυεί επιχειρήσει για να δημιουργούν νέα προϊόντα και να τα φέρνουν στην αγορά. Και ε, πράγματι σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, ε, δηλαδή μέχρι στιγμής ε, δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία με τις δημιουργικές ε, μέσα στο δημιουργικό τομέα. Αλλά από εκεί και μετά και στις δημιουργικού στους δημιουργικούς κλάδους έχουμε για παράδειγμα εκείνον της ε, μουσική ή άλλων τεχνών που είναι κατακαιρματισμένοι μεταξύ του. Άρα λοιπόν το να φέρνουμε μέσα αυτής της πρωτοβουλίας ε, τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορεί σε επαφή μεταξύ του έχει πολύ ιδιαίτερο νόημα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κλίμακα την οποία μπορούμε να επιτύχουμε και το τι υπάρχει σε επίπεδο συνεργασία. Τώρα έρχομαι σε αυτό το ερώτημα που θέσατε κυρία Πρόεδρε προ το τι θα περιλαμβάνει το μελλοντικό Horizon. Ε, δεν είμαι εγώ αρμόδιο να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνα που σχεδιάζει το μελλοντικό πρόγραμμα και εκείνη θα αποφασίσει. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει μια χρωματοδότηση από το Horizon 2020 μέσω άλλων τρόπων ε, ή μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Εμείς ουσιαστικά εδώ καταδεικνύουμε με ποιον τρόπο προωθούμε την κοινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και μετά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα διαμορφωθεί η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας στο Horizon. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος, η Επιτροπή θέλει να τοποθετηθεί. Ανετικό νεύμα από την Επιτροπή. Οπότε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τομέα, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κέν, για τις τοποθετήσεις σας εδώ, για τα όσα μας ε, εξηγήσατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και σίγουρα αν το χρόνο θα σας ε, καλέσουμε και πάλι εδώ για να μας ε, ενημερώσετε σε σχέση με τα επιτέλματα αυτά που θα προκύψουν δηλαδή από τις νέες πρωτοβουλίες σας στον χώρο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ja. Wir sind hier vorne gerade. Ναι, έχουμε εκπλαχεί λίγο από την πλευρά του Προεδρείου για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε να κάνει κανένα σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτέ τι φήμε. Αλλά εντάξει, το κρατάμε αυτό. Έκπληκτη. Μεν, αλλά το σημειώνουμε. Φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή μα σα διάταξη. Ε, εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους ε, τους συναδέλφους της Επιτροπής και θα παρακαλέσω τους συντονιστές μας να παραμείνουν εδώ για την συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα ξεκινήσει σε περίπου 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.